Και το λόγο λοιπόν έχει ο Επίτροπος Άντζεπ. αλλά αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Επίτροπε, θα περιμένετε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ομιλία του Επιτρόπου Άνση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πολύ μεγάλη μια πρόοδο για τη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής αγοράς για την Ευρώπη με δύο δέσμες μέτρων ε, και πρωτοβουλειών. Το πρώτο αφορά το διασυνοριακό ε, διαδικτυακό εμπόριο στην Ευρώπη που άρει τα εμπόρια, αυξάνει, εμπόδια, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών και δημιουργεί κατάλληλο ε, ε, πεδίο ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Το δεύτερο αφορά την δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακές πλατφόρμες και μέσα μετάδοσης. Και τα δύο είναι δεσμεύσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, στρατηγική για την ψηφιακή ενία αγορά, την οποία παρουσίασα εδώ στο, ε, στο Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, πριν από ένα χρόνο και τα δύο αφορούν την αγαστή λειτουργία της ψηφιακής ενίας αγοράς σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς ε, θα ήθελα να αναφερθώ στη δέσμη μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου ώστε να γίνει πραγματικά πανευρωπαϊκή με ισότιμους όρους ε, για τους καταναλωτές ε, και τους εμπόρους σε όλα τα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ανταλλαγή περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών πλέον από το διαδίκτυο και αυξάνεται συνεχώς ε, η κίνηση. Επομένως ε, ε, θα πρέπει να αλλάξουμε και την αργή κίνηση της νομοθεσίας. Οι καταναλωτές αξίζουν περισσότερα, δεν μπορούν να περιορίζονται μόνο στην εσωτερική τους αγορά πρέπει να μπορούν να εκμεταλλεύονται και τις δυνατότητες που προσφέρονται από την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφιακή εποχή η δέσμη μέτρων αφορά τρεις βασικά τομείς. Πρώτον, δεν θα επιτρέπει άδικες διακρίσεις και διαδικτυακά αλλά και εκτός δικτύου. Σε μια πραγματική ενιαία αγορά δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση ε, λόγω της εθνικότητας, ε, της κατοικίας ε, ή της χώρας διαμονής κάποιου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πουλούν και να παραδίδουν αγαθά σε όλες τις ευρωπαϊκές αγοράς. Εάν ένας καταναλωτής όμως πηγαίνει σε ένα διαδικτυακό κατάστημα θα πρέπει να την χάνει της ίδιας μεταχείρισης με τους ημεδαπούς και δεν θα πρέπει να παρακολύεται η υποχρέωση να παραδίδεται το αγαθό. Οι έμποροι θα πρέπει να μην έχουν κανένα εμπόδιο και θα πρέπει να παραδίδουν τα αγαθά όπως ε, θα τα παρέδιδαν σε κάποιον από τη χώρα τους. Δεύτερον, θα αυξηθεί η διαφάνεια των ε, τιμών παραίδευσης, ε, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα επιτρέπει ανταγωνισμό μεταξύ ε, των διαφορών χωρών διασυνοριακά. Αυτό θα βοηθήσει τους καταναλωτές ε, να έχουν καλύτερες προσφορές και επίσης μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογές θα βοηθήσει περισσότερους λιανοπολιτές ε, διαδικτυακά να προσεγγίσουν περισσότερο τους πελάτες και ε, θα επιτρέπει σε περισσότερους παρόχους διαδικτύου ε, να δραστηριοποιούνται. Και φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιβάλλεται μία τιμή σε όλη την Ευρώπη. Τρίτον, η δέσμη μέτρων μας θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων στο διαδικτυακό εμπόριο, θα μειώσει τις αθέμητες πρακτικές και θα αυξήσει τα δικαιώματα των καταναλωτών διασυνοριακά. επιπλέον θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ε, εθνικών ε, αρχών προστασίας των καταναλωτών. Ο στόχος είναι να άρουμε τα βασικά εμπόδια για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, οι διαδικτυακές πλατφόρμες είναι μια νέα πραγματικότητα στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει και να τις υποδεχτεί αυτές τις πλατφόρμες έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε, πουλάμε και εμπορευόμαστε και πώς διασκεδάζουμε, διαβάζουμε, μελετούμε. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη για τους καταναλωτές, για την ευρύτερη κοινωνία, για την ε, βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η βασική αρχή και ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες ε, προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει καινοτομία ε, ε, εκ των άνω και επίσης θα πρέπει να γίνεται με ανοιχτό και δίκαιο τρόπο. Αυτό σημαίνει ισότιμες συνθήκες για θεμητό ε, και ανοιχτό ανταγωνισμό. Οποιοςδήποτε συμμετέχει στην αγορά, είτε σε παραδοσιακό ε, μέσο είτε διαδικτυακά, θα πρέπει να μπορεί να ε, δραστηριοποιείται χωρίς διακρίσεις. Οι πλατφόρμες είναι καινοτόμες και έχουν θετικές συνέπειες για την οικονομία μας και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, όπως καταδεικνύεται από τις μελέτες. Καταδεικνύεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά καλή σε τομεί όπως η οικονομία των εφαρμογών, ε, τα οικονομικά και τη συνεργατική οικονομία. Προκειμένου να μπορέσουν λοιπόν να ανθίσουν όλες αυτές οι πλατφόρμες και οι ευρωπαϊκές, ε, χρειάζεται ένα κατάλληλο νομικό περιβάλλον που θα τους προσφέρει ασφάλεια δικαίου. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε απόλυτα σαφείς στην ανακοίνωσή μας δεν θα υπάρχει κανένας νέος οριζόντιος κανονισμός ή ρυθμιστής για τις πλατφόρμες. Δεν θα αλλάξουμε το παρόν πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ε, διατάξεις ε, περί ευθύνης. Βεβαίως οι πλατφόρμες αυτές, όπως και ο οποιοδήποτε άλλος ε, πάροχος του διαδικτύου ή η ενδιάμεση, πρέπει να σέβονται το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει επίσης να ε, δρουν υπεύθυνα όσον αφορά το περιεχόμενο και να υπάρχει διαφάνεια ως προς τις δραστηριότητές τους. Πρόκειται για σημαντικές αρχές. Γι' αυτό και έχουμε μια προσέγγιση με βάση τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε, που σημαίνει ότι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις πλατφόρμες όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, θα επιλύεται ε, βάσει των ε, κανόνων μας. Εάν υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά τις τηλεπικοινωνίες, θα επιλύεται βάσει των κανόνων τηλεπικοινωνιών. Τα πρώτα βήματα ε, προς αυτή την κατεύθυνση ελήφθησαν ήδη από σήμερα με την πρόταση που κάναμε για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τη σχετική οδηγία. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή αυτού του μέσου. Οι αρχές που ανέφερα φυσικά αφορούν και τις μεταδόσεις όπου πλέον υπάρχει σημαντική παρουσία διαδικτυακής παρουσίας και πλατφόρμες ε, και video on demand και πρέπει να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρούν τους ίδιους κανόνες. Επειδή ε, έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε την αρχή της χώρας καταγωγής. Οι υπάροχοι θα υπόκεινται στους κανόνες της χώρας στην οποία εδρεύουν. Η πρότασή μας ε, θα προσδώσει επίσης ευελιξία στους κανόνες διαφήμισης και θα δώσει όθηση στις προσπάθειές μας για να υπάρξει συνεργατική ευρωπαϊκή ε, εργασία. Θα προστατεύει επίσης τους ανηλίκους ε, που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να βλέπουν περιεχόμενο και θα υπάρχει και ε, ε, ρύθμιση από τους ρυθμιστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προσβλέπω στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις δύο σημαντικές ε, δέσμες μέτρων προτάσεων πραγματικότητα. θέλουμε να δημιουργήσουμε την ψηφιακή νέα αγορά που χρειάζεται η Ευρώπη, μια ψηφιακή αγορά όπου όλοι θα είναι κερδισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Το πάμε στους υποσχόμενους πολιτικών ομάδων. Πρώτα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον λόγο ο κύριος Ανδρέας Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, καταρχά, κύριε Αντιπρόεδρε, Άντσιπ, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και να σα συγχαρώ από πλευρά του ΕΛΚ για το πακέτο αυτό. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο έκανε με τόλμη τα απαραίτητα βήματα τα οποία έπρεπε να γίνουν και εκ παραλλήλου επέδειξε ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς εκείνους που πραγματικά χρειαζόμασταν πιο πολλές ε, πληροφορίε από τις αγορές για να είμαστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσουμε το σωστό δρόμο. Το βασικό που θέτεται είναι το, η πρόταση για τον γεωποκλεισμό. Γιατί δημιουργήθηκε ένας νέος κλάδος τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αγορά. Το παράδειγμα της Disneyland το Παρίσι ήταν το πιο εντυπωσιακό, αλλά υπάρχουν και άλλες διαπαθές όπου πραγματικά χρειάζεται ενότητα και ενιαίος χαρακτήρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε την κριτική σε ό,τι αφορά τους τομείς αυτούς και σε κάποιους τομείς θεωρούν κάποιοι ότι θα μπορούσαν να γίνουν πιο πολλά, αλλά Θέλουμε να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μα, προκειμένου στο τελική ανάλυση να υποφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε από το πακέτο αυτό. Είπατε ότι στι πλατφόρμε ε, θέλετε να επιβάλλετε μια οριζόντια ρύθμιση. Αυτό βάσει τη έκθεση και τη έρευνα του τομέα. Είναι σωστό αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας των πληροφοριών έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα για την πλατφόρμα της νομοθεσίας και είπατε ότι όπου υπάρχει ανάγκη θα γίνουν περαιτέρω βήματα ανά τομέα. Εμείς ως ΕΛΚ θέλουμε να υποστηρίξουμε την προσέγγιση αυτή γιατί πιστεύουμε ότι ο ευρωπαϊκός δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των πλατφόρμων online στην Ευρώπη αλλά και εκτός ε, Ευρώπης που συνεργάζονται εκτός Ευρώπης είναι κάτι το απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε την τελική ανάλυση ότι η νέα αγορά με 500 εκατομμύρια κατανάλωτες θα έχει ωφέλη για όλου. Και γι' αυτό λοιπόν είμαστε στις φάσεις διαβουλεύσεων από τη φάση και σας ευχαριστώ πολύ. Per ε, il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici, la parola... Η κυρία Γκέμπχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Άντσιξ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονό ότι μας παρουσιάσατε εδώ σήμερα το πακέτο αυτό, τα μέτρα τα, αυτά τα οποία προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πήρε καιρό, αλλά επιτέλους τα έχουμε, σας συγχαίρω. Λοιπόν και το κοινοβούλιο μας από το 2011 εργάζεται για την δρομολόγηση των μέτρων αυτών. Νομίζω ότι στον αναλογικό κόσμο θα ήταν πραγματικά αδιανόητο ένας πολιτής να ένας μάλλον ε, αγοραστής ε, και ένας καταναλωτής να μην γίνεται εκτός απαιτήσει σε ένα άλλο κράτος μέλο. μέλος. Τέτοια είδου πράγματα θα πρέπει να αποτρέψουμε με τη ρυθμίση για τον υγεία Αποκλείσμα, γιατί μιλάμε για τη δική μεταχείριση του κόσμου λόγω της χώρας στην οποία ζει ή λόγω της πιστοτικής κάρτας που έχει. Είναι απαράδεκτο αυτό σε μια ενιαία αγορά. Σε μια ενιαία αγορά όπου στο επίκεντρο θέλουμε να θέσουμε τον άνθρωπο. Μας είπατε ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλετε να ακολουθήσετε οριζόντια προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες. Συγχαρητήρια. Ήδη στην έκθεση του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο αναφέραμε ότι αυτό θα αποτελούσε εσφαλμένη προσέγγιση γιατί είναι τόσο διαφορετική διαμόρφωση όλων των πλατφόρμων αυτών που δεν μπορεί να υπάρξει μια λύση για όλους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά και προβλήματα του κάθε τομέα και ενδεχομένω να υπάρχει και τομεακή προσέγγιση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ο σωστό τρόπο να προχωρήσουμε. Και αυτό που επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το οποίο ελπίζω να γίνει στο πακέτο αυτό προς όφελος του καταναλωτή είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά το διαδικτύο για να μην είναι αδιαφανείς ε, οι πληροφορίες που δίδονται στον ε, καταναλωτή, να μην είναι κρυφά κάποια τέλη που επιβάλλονται ή μόνο στο τέλος μιας παραγγελίας, για παράδειγμα, να ανακαλύπτει ο καταναλωτή ότι δεν μπορεί να του στείλουν το πακέτο του γιατί είναι υπερβολικά υψηλά τα έξοδα αποστολής. Και επίσης ε, το θέμα είναι επίση να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο η αποστολή των πακέτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε πραγματικά να υπάρχει ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Τώρα για του VCR, το λόγο έχει ο κύριο Φέγκελ. Κύριε Επίτροπε, όλη μου τη ζωή ε, την έχω περάσει σε αυτόν τον κλάδο και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η Ευρώπη και στο σημείο αυτό και στον κλάδο αυτό κάνει όλα ε, βήματα προς τα πίσω και θα καταρρεύσει. Θα θυμάστε ε, που είχαμε την Expo, Bull, ε, η Ιταλία, η Βρετανία, την ICL. Ε, όλα αυτά πλέον είναι παρελθόν μακρινό. Όλα στην Αμερική και στην Ασία κρίνονται. Ένας λόγος γι' αυτό είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε ψηφιακή ενιαία αγορά. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Επιτροπής αυτής χωρίς αμφιβολία και παρά το γεγονός ότι η ομάδα μας έχει την άποψη ότι σε πολλά ζητήματα είναι υπερβολικά μεγάλη η παρουσία της Ευρώπης, θεωρώ ότι εδώ πέρα χρειάζεται ε, ευρωπαϊκή διάσταση. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε τις εργασίες σας. Για τους φιλελευθέρους τώρα. Έχει το λόγο η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε για κύριε Αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστούμε διότι διατυπώσατε αυτή την ε, καινούργια νομοθετική πρόταση και τι σχετικέ ε, ανακοινώσει. Θα πρέπει να σα πω ε, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και παρακαλώ να πιέσετε προ κάθε κατεύθυνση και κυρίω προ το Συμβούλιο, τόσο ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδρομή αυτή για την ε, ψηφιακή αγορά. Έχουμε αυτή την ε, πρόταση που πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή τη βδομάδα. Να αποδειχθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να γίνει πρωτοπόρα η Ευρώπη όσον αφορά την ψηφιακή επανάσταση. Πάντω, κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει να σα πω ότι ε, δεν αρέσουν σε όλους αυτές οι προτάσεις σας. Σπασότσο όχι όλους. Όσον αφορά τι ψηφιακέ συμβάσει, παρακαλώ να ολοκληρώσετε την προσπάθειά σας στο συνομότερο δυνατόν, τόσο ώστε ε, τα θέματα που έχουν μπλοκαριστεί να ξεμπλοκαριστούν τώρα. Επίση έχουμε και μια πρόταση που θέλουμε να έχουμε αυτού του είδους τα αγραία συστήματα επαλήθευσης, ούτως ώστε να μπορούν οι, οι χρήστες να παρακολουθήσουν κάποια ταινία. Ε, και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το αδικαιολόγητο γεωαποκλεισμό για του πολίτε. και θα πρέπει επίση να συνδυαστεί η προσπαθειά σα με περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή των δεμάτων θα πρέπει να υπάρχει επομένω εμπιστοσύνη από πλευρά ε, καταναλωτών αλλά και συναλλασσομένων γενικότερα ε, αυτό είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο οπότε θα πρέπει να προχωρήσετε για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση για την πλατφόρμα που είναι κάτι το τόσο ευρύ που σχεδόν καλύπτει τα πάντα. Οπότε προσοχή να μην έχουμε τελικά υπερβολική πανέβαση στην αγορά πλευρά νομοθεσία. Ευχαριστούμε. Πρόεδρο. Για τη συνοσπονδιακή άμαρα τη ε, Ευρωπαϊκή Συνοτική Αριστερά, ο κύριο Ντιγιόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εναρμονίσει όλου του κανόνε για τι ε, επιγραμμικές πωλήσει και να δημιουργήσει ε, τις ε, πωλήσει αυτές. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία όμως δεν θα επιληθούν σε κάποιες περιπτώσεις για τον καταναλωτέ. Δύο παραδείγματα να δώσω, αν και υπάρχουν πολλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να προβληθούν σε μηχανές αναζήτησης, σε Google, σε ε, μηχανές αναζήτησης και σύγκρισης ε, τιμών. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πιο πολλά λεφτά για να προβληθούν και το αποτέλεσμα είναι ότι ο καταναλωτή τελικά δεν έχει σωστή επισκόπηση όλων των παρόχων. Και αυτό που είναι πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα το μελετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δίνει κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αυτορύθμιση. Είναι μια απώλεια αυτό γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που έχουμε. Ζητώ να υπάρχει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον τομέα αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα, ένα πρακτικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν συχνά οι καταναλωτέ, οι τιμέ για τις, τα εισιτήρια για συναυλίε. Υπάρχουν τέτοια ιστοσελίδε που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουν τις ίδιες τιμές. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διαφορά που υπάρχει στις τιμές διαφορών παρόχων και για το πέρα δεν υπάρχει διαφάνεια. Και έτσι λοιπόν μπορεί να έχουν ξεπουληθεί ε, κάποια εισιτήρια στην επίσημη στο σελίδα, αλλά να διατύφονται τα εισιτήρια αυτά σε άλλες τιμές από άλλους παρόχους. Θα το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Ρέντα για τους πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η πρόταση κανονισμού για το geo-blocking ε, θα μπορούσε να είναι ε, πολύ καλή αν είχατε υπάρξει λίγο πιο φιλόδοξη. Υπάρχουν καλοί λόγοι για να προχωρήσουμε την πρόταση αυτή, ε, έχει καλά στοιχεία ε, αντιμετωπίζει τις ανησυχίες ε, του νομοθέτη, αλλά ταυτόχρονα χάνει και την ουσία του προβλήματος. Ξέρουμε όλοι ότι όταν γνωράμε, ε, ρωτάμε τους καταναλωτές τι άποψη έχουν για το geo-blocking, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι αυτό το βίντεο δεν διατίθεται στη χώρα σας. Βεβαίως τα βίντεο εξαιρούνται τελείως από τον κανονισμό και από ό,τι φαίνεται την τελευταία στιγμή και άλλο περιεχόμενο το οποίο ε, καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογή. Είπατε ότι θα ρυθμίσουμε αυτό στις προτάσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά υπάρχει πολύ geoblocking ε, υλικού, κυρίως ε, ε, βίντεο υλικού, που δεν έχει καμία σχέση με πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται να το δει κάποιο σε άλλη χώρα. ελπίζω λοιπόν στα οπτικοακουστικά ζητήματα να αντιμετωπίσετε και το θέμα βίντεο που δεν αφορούν θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Πολύ συχνά μπορεί να είναι ο πολιτής αυτός ο οποίος αποφασίζει ότι για εμπορικούς λόγους θα του επιφέρει μεγαλύτερο κέρδος να χωρίσει την αγορά. Επομένως θα πρέπει να προσέξετε να μην δημιουργήσετε κανένα ρυθμιστικό κενό ώστε στο τέλος ε, πραγματικά να έχουμε το τέλος ε, του geo-blocking ε, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Για την Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Επιτροπέ. Αν σε πριν από ένα χρόνο περίπου μας παρουσιάσατε τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά που περιλαμβάνει διάφορα σημεία για την καλύτερη πρόσβαση για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές ε, για την καλύτερους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και είχατε πει τότε ότι πρόκειται για 11,7 δις ε, τα οποία θα μπορούσαν να γλιτώσουν οι καταναλωτές ανά έτος αν υπήρχε καλύτερο ηλεκτρονικό εμπόριο, ένα δεύτερο πακέτο ε, για την νέα αγορά επειδή ε, φυσικά όλα αυτά τα εμπόδια αποτρέπουν το λειτουργικό εμπόριο και όχι ο αποκλεισμό, όπου χρειαζόταν μια ισορροπία μεταξύ τη ε, ασφάλειας δικαίου και των συμφερόντων των καταναλωτών. Και το τελευταίο θέμα είναι καλύτερη πρόσβαση στα ψηφιακά περιεχόμενα. Θα πρέπει να σας, σας πω ότι το σημερινό πακέτο σίγουρα θα βελτιώσει την ασφάλεια του καταναλωτή, θα βελτιώσει και το online shopping και θα είναι πιο ευνοϊκό για τον καταναλωτή. Το κατά πόσο θα είναι ικανοποιημένος ο καταναλωτής ε, δεν το ξέρουμε, αλλά εν γέννη πρόκειται για μια βελτίωση και θέματα εμπιστοσύνης βελτιώνονται σε ό,τι αφορά τις αβετιότητες σε ό,τι αφορά την καλύτερη ταυτοποίηση και φυσικά και τα εθνικοί προπολογισμοί θα είναι πιο ε, πλήρη σε ό,τι αφορά το 20% του οπτικοακουστικού κλάδου που είναι ευρωπαϊκής προέλευσης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και φυσικά θα είναι ευχαριστημένα και τα πολιτισμικά μέσα. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επιτροπέ. Παλιά το να αγοράσει κανείς ένα αγαθό σήμαινε να πάει στο μαγαζί, να δώσει χρήματα και να επιλέξει τι ήθελε να επιλέξει και μετά να επιστρέψει ήσυχο ήσυχο στο σπίτι τους. Έτσι ψωνίζαμε εμείς ως παιδιά. Φυσικά άλλαξε από τότε ο κόσμος. Και ιδιαίτερα ε, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Σήμερα λοιπόν, συχνά δεν πηγαίνουμε οι ίδιοι στα μαγαζιά για να αγοράσουμε ένα προϊόν. Όχι, καθόμαστε στον υπολογιστή μας, στην ταμπλέτα μας, μη σας πω και στο κινητό μας και αγοράζουμε έτσι προϊόντα από το διαδικτύο. Και πού λοιπόν προκύπτει το πρόβλημα. Προκύπτει στο ότι τα αγαθά δεν βρίσκονται πλέον ε, κοντά μας, αλλά κάπου αλλού στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι η τεχνολογία μας διευκολύνει προς την κατεύθυνση αυτή στο να επιλέξουμε τα προϊόντα, αλλά η πληθώρα των κανόνων που είναι διακριτική, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή και τελικά εξαρτάται από το που βρίσκεται ο καταναλωτή, σε ποια χώρα Ω προ αυτά λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πάρα πολλοί διαφορετικοί παράγοντε όπω είναι οι τιμέ, ή ο τόπο στον οποίο βρίσκεται κανεί. Και προ την κατεύθυνση λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα του για αποκλεισμό. Γιατί η ενιαία ψηφιακή αγορά θα πρέπει να οικοδομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ακριβώ με τον ίδιο τρόπο όπω ε, δούλευε παλιά το να πάει κανεί στο μαγαζί. Ευχαριστώ κύριε Κάρινς. και κυρία Τόγια. Σήμερα η ανάπτυξη, αντίθετα με το παρελθόν, θεμελιώνεται σε δύο βασικά στοιχεία, στην ενέργεια, στην ενέργεια και στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αν θέλουμε να έχουμε βιωσιμότητα και παγκόσμια διάσταση, λοιπόν. Γι' αυτό, κύριε Επίτροπε, εκτιμούμε ιδιαίτερα την ενιαία ψηφιακή αγορά, τα μέτρα τα οποία ξεκινούν και όλες τις συνδεδεμένες υπηρεσίες, γιατί είναι η νέα αρχιτεκτονική δομή, είναι οι κανόνες, τα νέα δικαιώματα αυτού του κόσμου που πλέον αναπτύσσεται σιγά-σιγά. Ε, ελεύθερη πρόσβεση, χωρίς φραγμούς, ε, σίγουρα θα δώσει μεγαλύτερες ευκαιρίες. Και πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα που πολίτες και επιχειρήσεις, καταναλωτές και πάροχοι μπορούν να κάνουν από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονό ότι μπορούν να έχουν φορητότητα των δικαιώματων τους ε, ψηφιακά, δικαιώματα κατανάλωσης, δικαιώματα και αξίες θα μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς όρια και εμπόδια και ακόμα και μικρές επιχειρήσεις που σήμερα φοβούνται πάρα πολύ αυτές τις αλλαγές, εμπορικέ και παραγωγικές επιχειρήσεις, θα πρέπει ε, να τις βοηθήσουμε να περάσουν ε, στην ψηφιακή εποχή. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την νομοθεσία. Ακούστηκε και από τις διάφορες παρεμβάσεις. Θα εξαρτηθεί από την νομοθεσία το πώς θα διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία χωρίς κινδύνους. Σαφής, ευέλικτη νομοθεσία που θα προσέχει όλα τα δικαιώματα και τα οικονομικά και τα παραγωγικά αλλά και την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια με κάθε έννοια και τα νέα δικαιώματα και προσωπικά και συλλογικά. Εμείς ε, αναφερόμαστε σε υπηρεσίες, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε, γιατί εγώ είμαι και από την Επιτροπή Βιομηχανίας, δεν μπορούμε λοιπόν να λησμονούμε ότι ε, η ψηφιακή τεχνολογία επενδύει σε όλο τον παραγωγικό κόσμο μαζικά ο παραγωγικός τομέας και οι υπηρεσίες αναμειγνέονται. Αναμειγνέονται και στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων αλλά και στις παραγωγικές διαδικασίες, στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και στις νέες ε, βιομηχανικές σχέσεις. Το όλο θέμα της ε, βιομηχανίας 4.0. Και φυσικά μεγάλη σημασία θα έχουν και υποδομές. Χωρίς υποδομές δεν μπορούμε να έχουμε ευρυζωνική ανάπτυξη και ε, όσον αφορά την ανακατανομή των συχνοτήτων ε, θα πρέπει ε, να να δώσουμε στις προνομιούχες συχνότητες για την ανάπτυξη των υποδομών και των τηλεπικοινωνιών. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο αυτά, υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας και η εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τόγια, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Θέλετε να απαντήσετε. Ο Τζαμπάς και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Τόγια, αναφερθήκατε στη βιομηχανία, στους καταναλωτές. Δεν νομίζετε ότι αυτό είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και αυτό έπρεπε να έχουμε σε αυτή την πρόταση. Να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των συμφορώντων των επιχειρήσεων και των καταναλωτών χωρίς ε, να βαραίνει η πλάστικα προς καμία κατεύθυνση. Κύριε Τόγια, παρακαλώ. Μα εγώ αναφέρθηκα ακριβώς σε διασυνδεδεμένε διατάξεις, διότι πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά διάφορες παρεμβάσεις. Υπάρχει η πράξη για την ενία ψηφιακή αγορά, υπάρχει βιομηχανία 4.0, υπάρχουν όλες οι ε, διαδικασίες ε, που αφορούν ε, τις παραγωγικές διαδικασίες, το μεταπητικό τομέα. Δεν είναι τα πάντα σε αυτές τις νομοθετικές πράξεις, αλλά αναφέρθηκα σε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε συμπληρωματικά να αναπτύξουμε, γιατί εγώ βλέπω μια ολοκληρωμένη αγορά. Το εμπόριο, τη βιομηχανία, την ψηφιακή αγορά και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, γιατί η βιωσιμότητα είναι ουσιαστικός παράγον σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστούμε κυρία Τόγια. Η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να συνεργαστούμε σε όλη την Ευρώπη, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά θα συμβατεί με την ψηφιακή αγορά. Δεν θέλουμε να φρενάρουμε την ψηφιακή αγορά. Τόσο με την αποκλεισμό δεν θα πρέπει να ε, εξαναγκάζονται οι εμπορευόμενοι να ανοίξουν τις πόρτες σε όλες τις αγορές χωριστά όμω αυτό γίνεται και αυτό είναι ένα άχθος, ένα άχθος ιδίω για τις μικρότερες εταιρείε. οπότε αντί να έχει περισσότερη επιλογή ο καταναλωτής τότε γίνεται το αντίθετο τώρα να αφορά την πλατφόρμα θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω, να μην έχουμε γίνει νομοθεσία, αλλά μεγαλώνει η πλατφόρμα γιατί το θέλουν οι καταναλωτές. Άρα θέλουν περισσότερες πλατφόρμες και περισσότερο ανταγωνισμό σε αυτές. Τώρα όσον αφορά την ευθύνη του ενδιάμεσου. Αυτό ίσως για τις νεοφύς επιχειρήσεις είναι ένα πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά τα, νέα μίντια, αυτό το αρέσει στους αλλά δεν πρόκειται για το ίδιο όσο για αυτό που προσφέρεται από τους παραδοσιακούς παρόγους, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση. Ευχαριστώ. Ονορεύλε Κάλλας. Κάλλας. Σας ευχαριστώ. Ο Τόμας Έντισον είχε πει ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος. Βρείτε τον. Να, ε, αυτό πάει να πει ψηφιακή καινοτομία. Επίλυση προβλημάτων, ε, εμπορεύματα, περιβάλλον, κινητικότητα, όλα αυτά. Και η στατική την ενιαία αγορά επίσης αποσκοπεί στο να έρθουν κάποιοι φραγμοί εκείνοι που από απαρχαιωμένες πρακτικές και απαρχαιωμένη νομοθεσία δημιουργούνται. Εξυγχρονισμός επομένως της νομοθεσίας αυτό θα κάνει την Ευρώπη μια ε, καινοτόμο πρωτοπόρα δύναμη. Δύο την για τον γεωποκλεισμό. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για να καλύψουμε τον διαγωνισμό για τις εταιρείε και όσον αφορά τα δέματα και όσον αφορά τις ε, συμβάσεις, το copyright και το δίκαιο του καταναλωτή. Όσο υπάρχει για οι εταιρείε πρόκειται να συνεχίσουν τις ίδιες πρακτικές. Ο σκοπός είναι να πουλούν ε, από το ίντερνετ περισσότερο οι εταιρείε και όχι να τις αποτρέψουμε. Τώρα κάτι άλλο όσον αφορά τις ε, μεταφορές. Δεν συμφωνώ με το επιχείρημα ότι θα πρέπει να υπάρξει παρέκκληση, να υπάρξει εξαίρεση. Πολλές φορές τα σχετικά website χρησιμοποιούνται από όλους τους Ευρωπαίους και εδώ πολλέ φορέ υπάρχει ο αποκλεισμό και εδώ υπάρχει δυσμενή διάκριση για του καταναλωτέ ανάλογα με το σε ποια χώρα μένουν και τι διεύθυνση Ιντερνετ έχουν. Άρα η στατική θα πρέπει να σημαίνει να σπάσουν τα φράγματα και τα εμπόδια. Να συνεχίσουμε λοιπόν την ίδια ρότα. Ευχαριστούμε κυρία Κάλλας. Και τώρα η κυρία Λόπες Μπερμέχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι ότι μεγαλύτερη, σας υπενθυμίζω μάλλον κύριε Επίτροπε, ότι είναι πρώτα εργαζόμενοι και μετά καταναλωτέ οι Ευρωπαίοι. Γιατί χωρί ε, έναν αξιοπρεπή μισθό δεν μπορεί να καταναλώσει. Θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει μόνο μια ψηφιακή αγορά. Γιατί εδώ, όμω εδώ ε, κανεί ε, στρουθοκαμιλίζει και δεν λαμβάνει την υπόψη τι διαφοροποιήσει και τι επιπτώσει επίση στην εργασία. Γιατί για, όσον αφορά τα δέματα, εδώ προσοχή γιατί έτσι δυναμητίζουμε τα κρατικά ταχυδρομεία. Η σημερινή νομοθεσία έχει κάποια στοιχεία τα οποία προχωρούμε σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό είναι αδικαιολόγητο. Μια ανησυχεί το ότι θεωρούμε τις ε, πλατφόρμες, τις ε, θεωρούμε κάτι σαν νέα υπηρεσία. Όχι, δεν είναι έτσι και επίσης ένα οδηγός θα πρέπει να έχει ε, τα ίδια δικαιώματα είτε δουλεύει στο Uber είτε σε ένα άλλο ταξί. Τώρα όσον αφορά τις επικοινωνίες και τα ξενοδοχεία το θέμα δεν είναι να έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό σε σχέση με τις παραδοσιακές δομές αλλά θέλουμε να υπάρχουν και εδώ οι ίδιε υποχρεώσεις και δικαιώματα ε, για όλο τον τομέα. Ελπίζουμε ότι αυτό το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με την προηγούμενη ομιλητρία. Το θέμα αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο εμπρέως. Σωστό είναι να καταρτίζεται μια στρατηγική την ψηφιακή νέα αγορά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια ψηφιακή κοινωνία. Και αυτό λίγο μου λείπει από την πρόταση την οποία υποβάλλεται. Μιλήσαμε με τους δημοσιογράφους, με φοιτητέ ε, δημοσιογραφίας και με ρώτησαν ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τους είπα ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή δημοσιότητα. Αυτό χρειάζεται για μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Θέλουμε να καταργήσουμε τον αποκλεισμό για τα παιχνίδια, όχι όμως για τα βίντεο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς ε, κατευθύνονται όλα από την αγορά σε ό,τι αφορά και την πρόταση αυτή. Γιατί όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των παραγωγών, αν μπορούσαμε να θέσουμε μια ευρωπαϊκή συζήτηση Μιλάμε για ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει το διαδικτύο και δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό. Ο Επιτροπός Ούτσιγκερ δεν είναι μόνο για την ψηφιακή ε, οικονομία υπεύθυνο είναι και για την ψηφιακή αγορά και γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν στο πακέτο αυτό να το συμπληρώσουμε, να βάλουμε και άλλα στοιχεία. Για να μην βλέπουμε τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους μόνο ως καταναλωτές, αλλά και ως πολίτες, ως εκλογείς, ως μέλη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα τέτοιο πακέτο θα πρέπει να καταρτήσουμε. Κύριε Ρέιμον, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Θέλετε να απαντήσετε. Η κυρία Γιακονσάρη έχει το λόγο. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που είπατε. Και μιλάτε για ένα πρόβλημα αξιών σε ό,τι αφορά το πακέτο αυτό, σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο αυτό. Όχι μόνο δηλαδή για την τεχνική πτυχή. Έχω να ρωτήσω όμως το εξή. Έχετε σκεφτεί με τον τρόπο με τον οποίο η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου μας επιτρέπει να βελτιωνόμαστε σε βάση αυτών τους, τους ε, αλγόριθμους που προϋποθέτει η τεχνολογική εξέλιξη. Προσπάθησα πραγματικά σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό να τονίσω ότι το κριτήριο θα πρέπει να είναι η πιο ευρεία δυνατή δημοσιότητα και όχι να διαμορφωθεί το γεωποκλεισμό με τέτοιο τρόπο που να έχει τα μέγιστα ωφέλη για τις επιχειρήσεις και να τονιστεί μόνο η εμπορική διάσταση. Έγινε η συζήτηση αυτή και για την ουδετερότητα του δικτύου κτλ. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε ένα κερδοφόρο μοντέλο, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να θέσουμε την ε, μέγιστη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των καταναλωτών. Δεν είναι ακριβώ το ίδιο και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιλέγουμε πάντα την ε, δυνατότητα που θα επιτρέψει τη μεγίστη επικοινωνία για τους πολίτες μας. Σαφχάουζερ. Κύριε Επίτροπε, για άλλη μια φορά αναφέρεστε και πάλι σε άνοιγμα της αγοράς. Μια, ε, ένα άνοιγμα το οποίο θα πάει χωρίς όρια και θα αφήσει τα κράτη-μέλη υπό ξένη κυριαρχία δεν κάνετε τίποτα για τις ξένες τεχνολογίες που είναι οι τεχνολογίες που κυριαρχούν. Η ενιαία σας αγοράς κατά συνέπεια λοιπόν θα δώσει ακόμα περισσότερα ε, στοιχεία στην Google, στην Apple, στη Facebook. Θα συνεργαστεί με τις αμερικανικές υπηρεσίες για την Αμερική και τις επιχειρήσεις της κατά των δικών μας επιχειρήσεων. Εχθές ε, ε, είχαμε την πρώτη παγκόσμια πρώτη με την Αλκατέλ και η Γερμανία ήταν και αυτή σε ε, πολύ καλό επίπεδο. Θα πρέπει να ε, υπάρξει ένα ευρωπαϊκό μονοπόλιο και όχι η εσωτερική σας ανταγωνιστική κατάσταση και ε, δίνεται πράγματα υπέρ αμερικανικών και κινέζικων επιχειρήσεων γιατί δεν υπήρξε καμία προστασία για τις ευρωπαϊκές αγορές γιατί δεν είχαμε καμία προστασία και για τις εθνικές αγορές πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία και η Κίνα ε, κάνουν μια πολιτική για να αντιμετωπίσουν αυτές τις πρεκλώσεις, η Ευρώπη όχι. Σήμερα προτείνεται ένα ευρωπαϊκό νέφος. Εντάξει, αλλά ε, θα είναι εις βάρος των πολιτών που θέλουν να προστατεύσουν τα δεδομένα σας. Εσείς με την προσέγγιση σας μας κάνει να φοβόμαστε για το χειρότερο και σίγουρα θα ε, δημιουργήσετε προβλήματα σε εμά και θα τα δώσετε σε ξένες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Χωρίς πραγματική στρατηγική, ε, διότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν προστατεύουν την αγορά όπως κάνουν η Ρωσία και η Κίνα για να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Αυτό σημαίνει ότι υποκύπτουμε σε εξωτερικές δυνάμεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία φιλοδοξία γιατί δεν έχει όρια και δεν έχει κυριαρχία. Καταστρέφει στο όνομα του ανταγωνισμού και της ανοιχτή τάσης ε, τα κράτη που έχουν μια κάποια φιλοδοξία. Τη Γαλλία και τη Γερμανία δηλαδή. Είναι καιρός να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη με άλλα θεσμικά όργανα και να φύγουμε από εδώ. Κύριε Σαφχάουζερ, ε, υπάρχει πλεκάρτα για σας. Θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Χόκμαρτ. Άκουσα την παρέμβασή σας που αναφέρεται στο ρώσικο προστατευτισμό και στη ρωσική οικονομία και τον υπερασπίζεται. Όπως ξέρετε, η ρωσική οικονομία ε, δεν έχει ανταγωνισμό και κράτος δικαίου και γι' αυτό υποβαθμίζεται. Πώς μπορούμε να έχουμε ευημερία ε, στην Ρωσία που τη θεωρείται υπόδειγμα για σας. Πέστε μας για την ε, προστατευτισμό, την ανομία, τη λισταρχική αγορά που βλέπουμε στην Ρωσία. Πέστε μας ε, για τη Ρωσία και πέστε μας την ευημερία των Ρώσων που θα τη βρούμε. Η οποία υποβαθμίζεται κάθε χρόνο ε, και είναι ντροπή για σας να υπερασπίζεστε μια τέτοια χώρα. Έχετε το λόγο κύριε Σαφχάουσερ. Αγαπητέ συνάδελφε, θα πάρετε το πρώτο βραβείο καρικατούρας ε, στα όσα σας είπα. Τι σας είπα, σας είπα αγορές όπως η Κίνα και η Ρωσία κατάφεραν να προστατευτούν από την κυριαρχία των ΗΠΑ στις τεχνολογίες αυτές χάρη στην προστασία των αγορών τους. Είπα επίσης, και δεν πιστεύω ότι η Ρωσία αποτελεί υπόδειγμα, αλλά η Ρωσία είναι μια κυρίαρχη χώρα που έχει στρατηγική κυριαρχίας και έχει καταφέρει να ε, υπερασπιστεί τις βασικές ε, τεχνολογικές δοσμός της για την ε, προστασία της κοινωνίας της, των επιχειρήσεών τους και της δικής μας κυριαρχία. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φιλοδοξία και είναι πονίδιστο αυτό για την Ευρώπη. Θα ήθελα παρεπιπτόντως να σας δώσω μια καλή είδηση.